Ladies and gentlemen, perhaps everybody could take their seat. Κυρίες και κύριοι, καθίστε παρακαλώ. Ask these very nice gentlemen and gentlewomen. Αν έχετε την καλοσύνη οι φωτογράφοι να αφήσετε κάτω τις μηχανές σας ούτως ώστε να ξεκινήσουμε την ακρόαση. Two members still finding their seats. Έχουμε ένα-δύο συναδέλφους που ψάχνονται ακόμα να βρουν τη θέση τους. Um, welcome this evening to Mr. Καλώς ήσατε στην ακρόση του κ. Άνσιπ, υποψηφίου Αντιπροέδρου και Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ενία Ψηφική Αγορά. Καλωσορίζω τα μέλη της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών και της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας καθώς και τα πολλά μέλη της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Υποθέσεων Καταναλωτού, που είναι η καθήλυνα αρμόδια επιτροπή. Η ακρόαση έχει σαν στόχο να επιτρέψει στα μέλη να ζητήσουν, να απαντήσουν σε δύο ερωτήσει. Έχει τα προσόντα να είναι μέλος του Σώματος Ευρωπαϊκής Επιτροπή υποψήφιο και είναι ικανός να εκτελέσει τα συγκεκριμένα ε, καθήκοντα για τα οποία του είναι υποψήφιος. Σύμφωνα στις κατευθυντήριες γραμμές για την έξι Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογεί το Κοινοβούλιο τους υποψήφιους επιτρόπους βάσει των γενικών τους ικανοτήτων γνώσεων ευρω... προσωπικής ανεξαρτησίας και τις προσπάθειες που καταβάλουν για την επίτευξη ε, των ευρωπαϊκών στόχων και επίσης αν έχουν τις ε, ικανότητες και τα προσόντα ή συγκεκριμένα χαρτοφυλάκιο και τις δυνατότητες επικοινωνίας. Ο κύριος Σανσίπ απάντησε γραπτός σε προπαρασκευαστικό ερωτηματολόγιο και οι απαντήσεις έχουν διανεμηθεί σε όλα τα μέλη, σε όλες τις γλώσσες. Βέβαια είναι δημόσια αυτή η ακρόαση, μεταδίδεται στο διαδίκτυο Πολλοί έξω από αυτή την αίθουσα μας παρακολουθούν, τους καλωσορίζω και αυτούς. Να σας εξηγήσω ποια θα είναι η όλη δομή της ακρόασης. Θα μιλήσει αρχικά 15 λεπτά υποψήφιος επίτροπος και στο τέλος θα έχει ένα πεντάλεπτο στη διάθεσή του για να ολοκληρώσει την ε, όλη αυτή ακρόαση. Εν τω μεταξύ θα τεθούν 45 ερωτήσεις από ευρωβουλευτές ένα λεπτό για την ερώτηση θα διατίθεται και δύο λεπτά για την απάντηση. Και θα προσπαθήσω να σας κρατήσω όλους τα χρονικά περιθώρια που διατίθενται. Στο μέτρο του δυνατού είναι σημαντικό αυτό. Υπάρχει διερμηνία σε 23 ε, γλώσσες και όλοι οι ομιλητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα τους. Μου ζητήθηκε να σας υπενθυμίσω ότι για τους διερμηνείς σας παρακαλώ, αν έχετε την καλοσύνη να μην μιλάτε πολύ γρήγορα, ούτως ώστε να μπορούν να σας παρακολουθήσουν οι διερμηνείς. Αν έχετε την καλοσύνη να μιλάτε καθαρά, θα βοηθούσε πολύ. Και θα ήθελα να παρακαλέσω τον υποψήφιο επίτροπο, τον κύριο Άνσεπ, να προβεί στην αρχική